Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Θα ξεκινήσουμε τις εργασίες μας λοιπόν. Η ημερήσια διάταξη βρίσκεται στο φάκελο που έχετε μπροστά σας. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια και αντιρρήσεις, μπορεί να θεωρηθεί εγκεκριμένη η ημερήσια διάταξη. Σήμερα υπάρχει διερμηνία σε όλες τις ε, γλώσσες των μελών των Επιτροπών Ήτρε και Ένβη. Τα πρακτικά της συνεδριάσεως της Δευτέρας Δεκεμβρίου βρίσκονται επίσης στο φάκελό σας. Εάν μέχρι το τέλος της συνεδριάσεως δεν υπάρξουν παρατηρήσεις, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα και τα πρακτικά. Σήμερα έχουμε σημαντική ψηφοφορία. Βλέπω ότι είναι παρόντες και οι συνάδελφοι, αλλά και πολύ φιλοξενούμενοι. Πρόκειται εδώ για μια ψηφοφορία μακρά και δύσκολη Παρακαλώ λοιπόν όλοι να συνεργαστούμε. Αυτό σημαίνει ότι όταν ε, κάποιος αποφασίσει να μιλήσει ή να φύγει ή να το κάνει εν πάση περιπτώσει με τρόπο ε, ταχύ και χωρίς να προκαλεί πρόβλημα. Καλωσορίζω λοιπόν όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν έτσι ώστε να εκπονήσουν την έκθεση αυτή. Η συνεργασία ήταν πάρα πολύ καλή μεταξύ όλων όσων ε, εργάστηκαν και στην οργάνωση των εργασιών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο Γκρότ για την καλή συνεργασία ανάμεσα στις δύο επιτροπές ε, καθώς επίσης και τους εισηγητές Δελβό και Σιμάσκι. Ε, ξεκινήσαμε την διαδικασία ε, ε, κοινών επιτροπών. Οι εργασίες λοιπόν διεξήχθησαν από κοινού και για να διευκολυνθεί η διαδικασία οι επιτροπές συμφώνησαν οι πρόεδροι των επιτροπών να περιτροπής να προεδρεύουν. οι δύο πρόεδροι αποφάσισαν να χωρίσουν την, τον χρόνο της προεδρίας. Εγώ θα, θα είμαι πρόεδρος στο πρώτο τμήμα της ψηφοφορίας και ο συνάδελφος στο δεύτερο τμήμα. Σας παρακαλώ λοιπόν να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Εάν ο συνάδελφος Γκρότε θέλει να προσθέσει κάτι, παρακαλώ να το κάνει. Επιθυμώ και εγώ να σας ευχαριστήσω και εσάς και, όλες, και όλους τους συναδέλφους καθώς και τις γραμματείες που συνεργαστήκατε πραγματικά με στένος μέχρι τέλους. Ας αρχίσουμε λοιπόν και βλέπω ότι έχουμε ακόμα δύο εγγεγραμμένους. Λοιπόν, έχουν ζητήσει το λόγο και άλλοι συνάδελφοι, ο κ. Όπως είπατε έχουμε πάρα πολλές ψηφοφορίες. Η ομάδα μου δεν είναι τόσο ενωμένη όσο θα ήθελα και γι' αυτό θα ήθελα ανάμεσα στο τέλος της ε, ψηφοφορίας των τροπολογιών και της τελικής ψήφου πέντε λεπτά διάλειμμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα γι' αυτό. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μιλώ εξ ονόματος πολλών συναδέλφων. Ε, πρέπει να σας πω ότι τον κατάλογο ψηφοφορίας ε, τον ε, ε, πήραμε πάρα πολύ αργά ε, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Δεν είναι δυνατόν την τελευταία στιγμή να λαμβάνουμε έναν τόσο μακρύ κατάλογο ψηφοφορίας. Ε, ε, νομίζω ότι θα πρέπει η ψηφοφορία να μην λάβει χώρα, γιατί δεν είναι δυνατόν να βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση η οποία θα είναι σωστή και ε, με, με τα λόγου γνώσεως. Δεν είναι δυνατόν, δεν είχαμε το χρόνο και την δυνατότητα ε, από το πρωί που πήραμε τις, ε, τη λίστα των ψηφοφοριών να μελετήσουμε. Να την μελετήσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρόιλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνάδελφοι το έργο αυτό στο οποίο καταλήξαμε μέχρι τώρα ήταν μεγάλο, δύσκολο και χρειάστηκε να εκπονηθεί υπό μεγάλη πίεση χρόνου. Όσοι συμμετέσχουν, οι συγητές και οι συγητές και ιδίω οι συνεργάτες των γραμματιών και των επιτροπών και των ομάδων χρειάστηκε να δουλέψουν πολύ σκληρά ακόμη και στις χριστουγεννιάτικες διακοπές ακόμα και την πρωτοχρονιά. Δεν τα υποτιμώ όλα αυτά. Από την άλλη μεριά είναι αληθές ότι η χθεσινοβραδινή κατάληξη είναι απαράδεκτη. Δεν είναι δυνατόν βουλευτές να έρχονται εδώ να ψηφίσουν εκατοντάδες σελίδων και πάνω από 900 τροπολογίες χωρίς να έχουν την ευκαιρία πρώτα να τα διαβάσουν. Οι συνάδελφοι που διαματήθηκαν ως τώρα έχουν 100% δίκιο, διότι δεν έχουν παρά μια μονάχα δυνατότητα να ακολουθήσουν πιστά τις λίστες ψηφοφοριών των πολιτικών ομάδων. Αυτό δεν είναι έντιμο, δεν είναι ούτε και αντικειμενικά ορθό, διότι υπάρχουν και μέσα στις πολιτικές ομάδες και αποκλίνουσες απόψεις. Ειδικά για το θέμα αυτό δίστανται οι απόψεις και εντός των πολιτικών ομάδων. Εάν θέλει κανείς να εκφράσει άποψη ψηφίζοντας διαφορετικά κάποιες από τις τροπολογίες, πρέπει να έχει τη δυνατότητα. Δεν έχει όμως τη δυνατότητα όταν λαμβάνει νύχτα τις τροπολογίες. Με τα λόγια μου αυτά δεν απευθύνω μομφή προς τις και τους συναδέλφους και συνεργάτες οι οποίοι εργάστηκαν μέχρι τώρα και όπως είπα τόσο σκληρά. Είναι εκ της φύσεως του πράγματος και κλιμακώθηκε με τον τρόπο αυτό. Επειδή όμως κλιμακώθηκε με τον τρόπο αυτό, οφείλουμε να συναγάγουμε κάποια συμπεράσματα και να πούμε κάθε βουλευτής πρέπει να έχει την δυνατότητα να αξιολογήσει τα κείμενα. Δεν είναι δεδομένο καθόλου αυτό και θεωρώ την διαδικασία αυτή ότι δεν είναι δημοκρατική και έντιμη. Δελβό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όντως, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα συζητούμε γι' αυτό το εξαιρετική σημασία θέματα. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για το θέμα αυτό ε, και είχαμε πολλές ομάδες εργασίας και ελπίζω πραγματικά ότι αυτοί που θα ψηφίσουν σήμερα δεν ε, ανακαλύπτουν ε, σήμερα είναι υλικό εντελώς νέο. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι τις 2.30 το πρωί ε, έκανα ε, αυτήν την, ε, κατάρτισα αυτό τον κατάλογο ψηφοφορίας και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω και την γραμματεία. Δουλέψαμε πάρα πολύ με την γραμματεία και νομίζω ότι δεν είναι καθόλου ορθό να έρχονται σήμερα συνάδελφοι και να λένε δεν πρέπει να ψηφίσουμε, πρέπει να αναβληθεί η ψηφοφορία. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Η συνάδελφο όλου. Ευχαριστώ, λυπάμαι. Αλλά μιλάμε για μια ξεκάθαρη προσπάθεια κολυσιεργίας. Συμφωνώ με τον κύριο Ρόιλ ότι η γραμματεία, οι συνεργάτες και οι σύμβουλοι μας εργάστηκαν εξαιρετικά σκληρά κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών για την προετοιμασία των ψήφων θα ήταν ε, πραγματικά άχρηστο να ακυρώσουμε ή να αναβάλουμε την ψηφοφορία γιατί αυτό ακυρώνει την προσπάθεια που έγινε κατά τη διάρκεια των διακοπών. Ας προχωρήσουμε παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι δεν θα πρέπει να αναβάλουμε ψηφοφορίες. Πολύ συχνά όταν ψηφίζουμε στις επιτροπές υπάρχουν δυνάμεις που τίνουν στην αναβολή διότι δεν έχουμε δίθεν εμβαθύνει. Εμείς είχαμε συμφωνήσει να ψηφίσουμε σήμερα. Το συζητήσαμε κατά τη διάρκεια της τελευταίας μας συνάντησης ότι θα ψηφίζαμε την 9η Ιανουαρίου. Αυτό το χρήσιμο αποτέλεσμα λοιπόν ε, είναι καρπός της προσπάθειας των δύο επιτροπών μας. Πρέπει να δημοσιεύσει το κείμενό της Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Ιανουαρίου και δεν θα πρέπει εμείς να αρνηθούμε την επίδρασή μας στην διατύπωση της μελλοντική ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία σήμερα. Ευχαριστώ Έλερ. αμφισβητώ ιδιαίτερο στην επιχειρηματολογία της εισηγήτριας. Το θέμα εδώ είναι ότι τα δικαιώματα των ευρωβουλευτών περικόπτονται. Δεν έχει καμία σχέση με τον σεβασμό που οφείλουμε στην εργασία και των εισηγητών και των σκιωδών εισηγητών και των συνεργατών. Εδώ το θέμα είναι ότι οι ευρωβουλευτές πρέπει να γνωρίζουν, έχουν εικόνα του τι ψηφίζουν. Και ούτε είναι ορθό να ζητούν από τους ευρωβουλευτές να καθίσουν ξύπνη μέχρι τις 3 τη νύχτα για να διαβάσουν την έκθεση. Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια προσπάθεια μιας μικρής πολιτικής ομάδας να επιβάλλει απόψεις σε μια μεγάλη πολιτική ομάδα. Γι' αυτό και ζητώ να αναβληθεί η ψηφοφορία. Ο συνάδελφος Οντί. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ προσωπικά ε, νομίζω ότι οφείλω να ακολουθήσω την τοποθέτηση του συναδέλφου Ερμπέρ που εκπροσωπεί την ε, ομάδα μας, αλλά οφείλω να σημειώσω ότι για μία ακόμα φορά δεν έχουμε μετάφραση των συμβιβασμών στη γλώσσα μας. Ε, βλέπουμε ότι η πολυγλωσία υποφέρει όλο και περισσότερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίσης ότι εδώ πρόκειται για μία έκθεση πρωτοβουλίας πιστεύουμε ότι μπορούμε μέσω αυτής της εργασίας μας ε, να επηρεάσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ αναρωτιέμαι και έχω πολλές αμφιβολίες. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ενέργειας το οποίο θα συγκληθεί ε, την Άνοιξη και θα υπάρξουν ε, πολλά έγγραφα τα οποία θα υποβληθούν εκεί και το έγγραφο του Κοινοβουλίου και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η άποψη των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων που ε, θα ε, εισαχθούν κατά κάποιο τρόπο στην, ε, στα προεκλογικά κείμενα των ευρωεκλογών. Νομίζω ότι επί των θεμάτων αυτών, όχι μόνο εν ώψη του 2030 αλλά και εν ώψη της προεκλογικής εκστρατείας, τα κείμενα αυτά θα πρέπει να γίνουν γνωστά. Ναι, τώρα, ε, εάν δεν ολοκληρώσουμε την εργασία σήμερα, ε, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε, γιατί διαφορετικά δεν θα έχουμε και χρόνο. Yes, thank you very much, Madam Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν ξεκινήσαμε τη διαδικασία αυτή εδώ και λίγους μήνες γνωρίζαμε ότι θα ήταν πολύ αμφίροπη εντατική διαδικασία και θα διαφωνούσαμε σε πολλά θέματα. Θέλω παρόλα αυτά να συγχαρώ και τους δύο εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές για μια εξαιρετικά θα έλεγα δοτική αν θέλετε μεταξύ τους της διαπραγματεύσεις στάση. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στην ποιότητα των συμβιβαστικών τροπολογιών. Είδαμε ελάχιστες αλλαγές στις ε, λίστες ψηφοφορίας από χθε. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος ξαφνικά σήμερα να αρχίσουν ορισμένοι να παίζουν ε, πολιτικά παιχνίδια ε, τις τελευταίες στιγμής ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Ας, ας σταματήσουμε λοιπόν περαιτέρω περιττές συζητήσεις και ας αρχίσουμε παρακαλώ την ψηφοφορία το ταχύτερο δυνατόν. Λοιπόν, τελευταίος ομιλητή, Α, όχι, τέσσερι έχω. Παρακαλώ να είστε σύντομοι, Μακένα. Σαν συντονίστρια της ε, ομάδας μου για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ζητώ να ψηφίσουμε σήμερα. Το χρονοδιάγραμμα ήταν γνωστό ε, σε όλους τους συναδέλφους εδώ και πολλές εβδομάδες. Οι τροπολογίες ήταν διαθέσιμες, οι λίστες ήταν διαθέσιμες και όπως ε, είπε η συγγήτρια υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες και στο εσωτερικό των πολιτικών ομάδων και γι' αυτό ακριβώς θα συζητάμε τα θέματα αυτά και γι' αυτό λοιπόν Πρόεδρη, ζητώ και από τους δύο να συνεχίσετε στις ψηφοφορίες. Το θέμα του πολιτικού χρονοδιαγράμματος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει ακριβώς ε, να δούμε την ψηφοφορία σήμερα σαν αυτό που είναι. Δηλαδή μια πολιτική απόφαση, όχι μια τεχνική απόφαση. Ας συνεχίσουμε λοιπόν. Ευχαριστώ. Χρώτε. Ευχαριστώ. Οι τροπολογίες έχουν κατατεθεί ήδη από τις 2 Δεκεμβρίου. Δεν ξέρω εάν πρέπει να παραταθεί η προθεσμία ώστε να μπορέσει και ο τελευταίος συναδέλφος, να τις ε, αναγνώσει. Από τις 2 Δεκεμβρίου υπάρχουν οι τροπολογίες. Οι συμβιβαστικέ τροπολογίες δε και κυκλοφόρησαν και πριν από τα Χριστούγεννα. Έχουμε μια καλή συνήθεια, δηλαδή τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Last minute changes αυτό το πρότεινε ο εισηγητή της Ήτρε και την δέχτηκα και εγώ. Εάν ακολουθούσαμε πιστά το γράμμα του κανονισμού δεν θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμβαστικέ τροπολογίε. Νομίζω όμω ότι ήταν αλεχθή λέχθηκε. Θα πρέπει να αρχίσουμε την ψηφοφορία και οτιδήποτε άλλο σημαίνει κολυσιεργία. Ευχαριστώ. Με κάθε σεβασμό που σας οφείλω είμαι υποχρεωμένος να επιμείνω ώστε γνωρίζω μεν τις συμβαστικές τροπολογίες αλλά δεν μπόρεσα να τις διαβάσω όλες και αυτές αποτελούν και την στοιχειώδη βάση των όσων θα έπρεπε να γνωρίζουμε εμείς ως μέλη, ως ευρωβουλευτές. Δεν πολιτικό λόγο εδώ, απλώς σας δηλώνω καθαρά ότι δεν γνωρίζω τι θα ψηφίσω. Σέμπερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όλοι έχουν επενδύσει πολύ χρόνο και βέβαια οι τελευταίες συμβαστικές προτάσεις κατέληξαν στα χέρια μας με μεγάλη καθυστέρηση. Έχουμε όμως ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα αν θέλουμε να ασκήσουμε κάποια επιρροή ως Κοινοβούλιο στις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, νομίζω ότι θα σημάνει και μια δημοκρατική εντιμότητα να θέσουμε το αίτημα αναβολής σε ψηφοφορία για να δούμε αν θα ψηφίσουμε ή όχι. Νομίζω ότι αυτό είναι έντιμο απέναντι σε όλες τις πλευρές. Και όποιος εν τέλει έχει την πλειοψηφία θα έχει κερδίσει. Πρόεδρος, νομίζω ότι η τελευταία, ο τελευταίος εγγεγραμμένος είναι αυτός που έκανε και μία πρόταση προς την Προεδρία, με την οποία η Προεδρία συμφωνεί. Γι' αυτό πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, θα ήθελα να ζητήσω να γίνει μία διακρύβωση όσον αφορά ε, τη, τους παριστάμενους. Ε, όλοι λοιπόν να κάνουμε μια δοκιμαστική ε, ψηφοφορία έτσι ώστε να ξεκινήσουμε ομαλά και ωραία τον, τη νέα χρονιά έτσι όπως επιθυμούμε όλοι. Να ξεκινήσει λοιπόν η διαδικασία. είναι test vote. And then we have to Voilà, il est un ALDE de trop. C'est... ALDE. E basta. Voilà. Ok, la machine marche. Bene. Πολύ ωραία. Έγινε η επαλήθευση των παρουσιών. Έχουμε μία ψήφο άλντε παραπάνω. Ωραία, να ψηφίσουμε λοιπόν την πρόταση του συναδέλφου Ζίμπερ ως εξής. Ποιος θέλει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας και επομένως να ψηφίσουμε. Όσοι θα πρέπει να υπερψηφίσουν. Διαφορετικά όσοι θέλουν αναβολή της ψηφοφορίας θα πρέπει να καταψηφίσουν. Άρχεται η ψηφοφορία. votazioni chiuse πέρας της ψηφοφορίας 65 ε, υπέρ ε, της συνέχισης ψηφοφορίας 50 ε, κατά και επομένως συνεχίζουμε και ψηφίζουμε. Ξεκινάμε με il compromesso 1 Συμβιβασμός 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κομπρομίσο 2. Συμβιβασμός 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Κατά την άποψή μου πρέπει να ε, ε, κάνουμε επαλήθευση. Μάλλον έχει απορριφθεί αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Votazione chiusa. Πέρας της 66 υπέρ, 58, 50 κατά, μία, τέσσερις αποχές, εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στον συμβιβασμό 10. Συμβιβασμός 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβιβασμός 11 υπέρ. Κατά. Τι να σας πω, θα πρέπει πρώτα να κάνουμε κάποιες, ε, κάποιους ελέγχους, γιατί δεν καταλαβαίνω πώς ψηφίζουμε. Ε, συμβιβασμός 11, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 52 υπέρ 62 κατά, επομένως απερίφθη. Συμβιβασμός 12 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 13, όχι, συμβιβασμός 14. Συμβιβασμός 14 ντεβε, υπέρ. Κοιτάξτε, ήρεμα και ωραία. Συμβιβασμός 14 ντεβε, όχι, δεν είναι συμβιβασμός, είναι ΔΕΒΕ 14. Δεν είναι συμβιβασμός. ΔΕΒΕ 14. Υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Τροπολογία 20, συγγνώμη, 216. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονική επαλήθευση επί του 216, παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 70 ψήφοι υπέρ 44 κατά, επομένω ενεκρίθη. Τροπολογία 219 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2.17 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση από της τροπολογίας 2.17. Πέρας. απερίφθη 57 υπέρ 59 κατά συμβιβασμός 5 υπέρ κατά Νομίζω πως εγκρίνεται, αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβιβασμός 5. Πέρας της ψηφοφορίας. 66 υπέρ, 50 κατά, επομένως εγκρίνεται. Συμβιβασμός 7 υπέρ, κατά. Απερίφθη κατά την άποψή μου, παρόλα αυτά ας επαληθεύσουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. 50 προς 65 επομένως απερίφθη. Συμβιβασμός 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Ηλεκτρονική επαλήθευση του συμβιβασμού 8. Παρακαλώ. Πέρας. 54 ψήφοι υπέρ, 65 κατά, επομένως απερίφθη. Συμβιβασμός 9 υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. 65 υπέρ 48 κατά, επομένως εγκρίνεται. Θα περάσουμε τώρα στην τροπολογία 253. Τροπολογία 253. Στη σελίδα 12 του καταλόγου σας. Τροπολογία 253. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2.48 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση κατά την άποψή μου έχει απορριφθεί, αλλά να το ελέγξουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. 66 υπέρ 51 ψήφοι κατά, επομένως εγκρίνεται. Τροπολογία 2.52 πρώτο τμήμα. 2.52 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά ηλεκτρονική επαλήθευση δεν ψηφίζουν ε, οι ομάδες ε, από κοινού, επομένως... Ε. Λοιπόν, δεύτερο τμήμα της 252, πέρα της ψηφοφορίας, εγκρίνεται 72 ψήφοι υπέρ 48 κατά. Τρίτο τμήμα της τροπολογίας 252 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.37 και 2.46 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.37 και 2.46 μαζί ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας 61 ψήφοι υπέρ 56 κατά, επομένως εγκρίνονται. Τροπολογία 2.51 υπέρ κατά κατά την άποψή μου με την ίδια πλειοψηφία παρόλα αυτά να επαληθεύσουμε. πέρα της ψηφοφορία. 62 υπέρ 56 κατά επομένως εγκρίνεται. Τροπολογία 2.50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 2.50 παρακαλώ. Chiusa Πέρας της ψηφοφορίας 65 υπέρ 54 κατά εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 276 στη σελίδα 17. Υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Η ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 2.76 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 66 υπέρ 50 κατά, επομένως εγκρίνεται. Δύο πενήντα οκτώ. Δύο πενήντα Υπέρ. Α, έκανα λάθος, λέει η Πρόεδρος. Τροπολογία 258, σελίδα 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 262. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Τροπολογία 257. Υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 266 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 266 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 66 υπέρ, 51 ψήφι κατά εγκρίνεται. 2.70, τροπολογία 2.70 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Ηλεκτρονική επαλήθευση τις τροπολογίες 2.70, παρακαλώ. Πέρας. 59 ψήφοι υπέρ, 60 κατά, απερίφθη. Λοιπόν, να κάνουμε μια επαλήθευση παρακαλώ, επιτρέψτε μας δύο λεπτάκια. Ζήτησε κάποιος το λόγο? Sì, prego. Can I ask, can μπορούμε να ξαναψηφίσουμε παρακαλώ την τροπολογία 270 γιατί ε, ε, οι μηχανές μας είχαν κάποιο πρόβλημα εδώ. Όχι, αυτό δεν είναι δυνατόν. 2,75. 2,75 παρακαλώ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 308. Υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 308 παρακαλώ. Πέρας. 58 υπέρ 59 κατά επομένως απερίφθη με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 281 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ επί της τροπολογίας 281. Πέρας. 62 υπέρ 56 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 292 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και σε αυτήν θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Τροπολογία 292 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 79 ψήφοι υπέρ 37 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 282 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 302 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 302. Τροπολογία 302 ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. 67 υπέρ, 44 κατά, επομένως εγκρίνεται. Τροπολογία 293 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Sul 293, prego. Ηλεκτρονική λοιπόν επί της 293, πέρας της ψηφοφορίας. 59 υπέρ, 55 κατά, εγκρίνεται. 2,85 υπέρ. Κατά. Αποχές, απερίφθη. 2,91 Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση από τις 2.85 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 60 υπέρ 58 κατά εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση είναι πολύ κοντινή σφιχτή η ψηφοφορία. Άρχεται λοιπόν πέρας της ψηφοφορίας. 57 υπέρ, 54 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 280 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.16. 3.16. 3.16 σελίδα 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 306. Παρακαλώ. Είναι πιο εύκολο ε, να παρακολουθούμε εάν μας λέτε και τη σελίδα γιατί ε, ε, περνάμε πολλές τροπολογίες και δεν είναι πολύ εύκολο να τις παρακολουθούμε. Ωραία, σελίδα 25, τροπολογία 306. adopted. Okay. Ja. No, no, only Bian. Adopté, adopté. Oui. C'est già adottato questo. Voilà, trois, c'est bien, c'est fait. Pagina 25. Τροπολογία 25, τροπολογία 306 ενώ η προηγούμενη τροπολογία ήταν η 316 και ενεκρίθη. Τροπολογία 306. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 306. Πέρας. 69 υπέρ 50 κατά εγκρίνεται. 318 υπέρ. Κατά. Αποχές. Κατά την άποψή μου εγκρίνεται η τροπολογία αυτή, αλλά καλύτερα να κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 66 υπέρ 49 κατά εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογία 283 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 289 σελίδα 27, 289 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Πέρας. 61 ε, ψήφοι υπέρ, 56 κατά εγκρίνεται. Ε, ήταν η 289. Στην επόμενη σελίδα τώρα έχουμε την τροπολογία 296. Υπέρ, κατά, απεριφθεί. Ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 296 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 39 υπέρ 75 κατά επομένως απερίφθη. Τροπολογία 278 στην επόμενη σελίδα. 278 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. 54 ψήφοι υπέρ, 59 κατά, επομένως απερίφθη. Τροπολογία 287 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 305 υπέρ. Κατά. Αποχές. Τι να σας πω, πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας της ψηφοφορίας. 60 υπέρ, 60 κατά, επομένως απερίφθη. Τροπολογία 324. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβιβασμός... Α, θέλετε επαλήθευση επί της 324. Ωραία. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 324. Ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν επί της 324 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 24 ε, υπέρ, 93 ψήφοι κατά. Επομένως απερίφθη. Συμβιβασμός 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 349 στην ε, σελίδα 35. Ε, σελίδα 35, τροπολογία 349. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Επαναλαμβάνω. Σελίδα 35. Τροπολογία 349. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Επόμενη σελίδα. 354. 354 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 353 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Επί της 353. Πέρας. 67 υπέρ 51 κατά δεκτή. Η κυρία Ντελβό, να σημειώσω εδώ ότι υπάρχει ένα μικρό λάθος στη λίστα για το ΕΛΚΑ. Αντί συν πρέπει να τεθεί πλην. Μιλάω ε, για την λίστα του ΕΛΚ μόνο. Για τη συμβιβαστική 19. Καλώς. Περνάμε στην ψηφοφορία λοιπόν. Ποιοι είναι υπέρ. Τη συμβιβαστική 19 επαναλαμβάνει πρόεδρος. Κοιτάξτε υπάρχει μια σύγχυση. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τη συμβιβαστική 19. Ψηφίζουμε. Τέλος. 40 υπέρ 76 κατά απορρίπτεται. Στην 37 συμβιβαστική 20 και είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Bene. Καλώς. Συμβιβαστική τροπολογία, ή μάλλον τροπολογία 314. 314. Στη σελίδα 37. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 314. Τέλος. 53 υπέρ, 53 κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 17. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Στη σελίδα 42 τώρα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 380 388 στη 45. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Επαναλαμβάνω στη σελίδα 45 τροπολογία 388. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 400. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 400. Παρακαλώ ψηφίζουμε. 67 υπέρ 49 κατά δεκτή. 401 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 375 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 375 ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. 51 υπέρ. 65 κατά. Απορρίπτεται. 398. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Από κοινού η 377 και η 397. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 374. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 378 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 382 πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το πρώτο τμήμα τώρα της 82, 382. Τέλος. 51 υπέρ, 64 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 399 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 21. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην 53. Στη σελίδα 53 λοιπόν, τροπολογία 424, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 424 πρώτο τμήμα. Τέλος. 65 υπέρ, 48 κατά δεκτή. Δεύτερο τμήμα της 424. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. ...64 υπέρ 51 κατά. Σελίδα 55, τροπολογία 431. Υπέρ. Κατά. Αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 23. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Πάμε στην σελίδα 57. Στην 444. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος ζητήθηκε για την 444. Ψηφίζουμε. Τέλος. 65 υπέρ 53 κατά δεκτή. 452 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 25 υπέρ κατά δεκτή. Συμβιβαστική αλφα μικρό υπέρ κατά. Αναφέρομαι ε, στην τροπολογία συμβιβαστική αλφα μικρό υπέρ κατά αποχές μου φαίνεται ότι απερίφθη αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 25α μικρό. Τέλος της ψηφοφορίας. 54 υπέρ, 57 κατά, απερίφθη. Πάμε τώρα στην 28. Συμβιβαστική 28. Υπέρ. Κατά. Απερίφθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 28 ψηφίζουμε. «56 υπέ, 59 κατά απερίφθη». Συμβιβαστική 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την συμβιβαστική 29. «57 υπέρ, 59 κατά απερίφη». Πηγαίνουμε τώρα στην 65. Μεγάλη ταχύτητα. 484. Υπέρ. Α, κάποιος έχει το λόγο. θα πρέπει να ψηφίσουμε και το 481 γιατί έχουν απορριφθεί όλες αυτές οι συμβαστικές. Μια στιγμή να επαληθεύσουμε. We Ζητάμε συγγνώμη, αλλά είναι περίπλοκα τα πράγματα. Ευχαριστώ τον Τούρμες. Βρισκόμαστε στη σελίδα 63. Τροπολογία 481. Η Πιλάρα έχει στο λόγο, αλλά χωρίς μικρόφωνο. Γιατί, Πρόεδρε, λέει ότι εκπίπτει ή αν η 35α εγκριθεί. Α, όχι. Α, όχι, δεν εγκρίθηκε. 25, ε, 25. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, λέγει η Αντελκαστήριο. Υπήρξε κάποια σύγχυση και μπερδεύτηκα. Είναι κατανοητό γιατί είναι περίπλοκη η ψηφοφορία. Ας περάσουμε τώρα στην σελίδα 63, τροπολογία 481 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το 481. Τέλος της ψηφοφορίας. 43 υπέρ 69 κατά. Siamo adesso a 64. Λοιπόν, στη σελίδα 64 τροπολογία 388 υπέρ επαναλαμβάνω είμαστε στη σελίδα 64 Α, για κάποιους άλλους είναι 63. Λοιπόν, ή στην 63 ή στην 64, όπου επιθυμείτε. Η τροπολογία πάντως παραμένει 488 είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 488. Πέρας της ψηφοφορίας. 53 υπέρ 55 κατά. Απορρίπτεται η 488. 483 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 484 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 485 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 480 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 480. Τέλος. 66 υπέρ, 46 κατά δεκτή. 477 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 477. Τέλος. 41 υπέρ, 69 κατά, απορρίπτεται. 482 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 482. Ψηφίζουμε. Τέλος. 39 υπέρ, 72 κατά απορρίπτεται. 298 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 298, ψηφίζουμε. Τέλος. 54 υπέρ, 55 κατά, απορρίπτεται. Από κοινού τώρα η 312 δεύτερο τμήμα και η 319 δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 848, επαναλαμβάνω, 848 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 848 ψηφίζουμε. Τέλος. 51 υπέρ, 53 κατά, απορρίπτεται. 476 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος. 52 υπέρ, 50 κατά, δεκτή. Συμβιβαστική 30 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 498 ενενήντα υπέρ. Στην σελίδα 69 για μένα λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω το 433 παράγραφος 2 πρέπει να ψηφιστεί ξεχωριστά ως προστίκη στην συμβαστική 21. No, entrambi i segretariati mi dicono che... Η γραμματεία μου λέει ότι έχει ήδη καλυφθεί. Έχει λοιπόν καλυφθεί. Περνάμε λοιπόν τώρα στην 488 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 488 Τέλος. 61 υπέρ 40 κατά. Δεκτή. 508 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 509 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 505 υπέρ κατά δεκτή 507 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα λοιπόν. Ψηφίζουμε. Τέλος. 54 υπέρ, 54 κατά, απερίφθη. Τροπολογία 503. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 502. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 503. Ψηφίζουμε. Τέλος. 55 υπέρ 52 κατά Τροπολογία 502 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 502. 54 υπέρ, 54 κατά, απερίφθη. 500 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 506 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 504 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος στην 504 τέλος 51 υπέρ 56 κατά απερίφθη Περνώ τώρα στον συνάδελφο συμπρόεδρο. Σας ευχαριστώ. Φτάσαμε στο ημίχρονο, πάρτε μια βαθιά ανάσα και συνεχίζουμε. Συμβαστική 33 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 735 υπέρ. Είναι στην επόμενη σελίδα στο δικό μου ε, έγγραφο. Ε. 735 υπέρ, λοιπόν, κατά, αποχές Επαλήθευση. 735 επαλήθευση. Τσεκ. Ψηφίσατε. Πέρας. Α, εγκρίνεται 104 ψήφους υπέρ. Δεν ε, μπορέσατε, δεν φάνηκε καθαρά ίσως επειδή πολλοί περιμέναν τη μετάφραση. 518 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 521 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 47 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 35. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, όπως και η συνάδελφό σας προηγουμένως, να μας ανακοινώνετε και τις σελίδες και τον αριθμό. Αν δεν λέτε τη σελίδα, σελίδα και αριθμό τροπολογίας, όπως έκανε η συνάδελφό σας συμπρόεδρος. Καλά, ας διαθέσουμε σε αυτούς τον απαραίτητο χρόνο. Λοιπόν, πρόκειται για την συμβαστική 35 σελίδα 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η επόμενη σελίδα 74 και είναι 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. «537» αυτή εκπίπτει. 538. Στη σελίδα 75 λέει ο πρόεδρος, ο διερμηνέας έχει μπροστά του σελίδα 76. Είναι άλλο εγγραφό. Στη δική μου περίπτωση ακούω τη μετάφραση μετά από την ψήφο. Δεν μπορώ έτσι να... Και εγώ λέει η κυρία Τελκαστήγιο και εγώ. Λοιπόν, πιο αργά παρακαλούμε, πιο αργά. Η 542 στη σελίδα 75-76. Υπέρ, κατά, Υπάρχει κάποιο πρόβλημα ακόμη, κυρία Χολ. Δεν ακούσαμε αγγλική μετάφραση για αυτό που είπατε κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κουάδρας, το πρόβλημα είναι διπλό. Αφενός πρόβλημα ταχύτητος. Αφετέρου δεν μεταφράζονται σωστά πάντα τα νούμερα. Ίσως αυτό οφείλεται στην ταχύτητα. Και το νούμερο που ακούμε από τη μετάφραση δεν αντιστοιχεί καμιά φορά. Καλά, α συνεχίσουμε. Ελπίζω από εδώ και μπρος όλα να είναι καλά. Βλέπω κάποιον ακόμα που ζητεί ε, το λόγο. Μήπως μπορείτε να λέτε καλύτερα 5-4-2 αντί 5-42 που στα γερμανικά είναι ανάποδα τα δύο τελευταία ψηφία. Μάλιστα, να λέω και τα νούμερα διαφορετικά. Καλά λοιπόν. Πού είμαστε τώρα 5-4-2 <laughs> αν με αυτόν τον τρόπο διευκολύνω τους συναδέλφους της Επιτροπής Βιομηχανίας να το κάνω. Ρέχα Τζέμπερ, εμείς αγαπούμε την πολυ, πολυγλωσία μας, αλλά κατ' εξαίρεση είναι αν θέλετε να μιλήσετε αγγλικά μπορείτε να διευκολύνετε όλους και όλους. Καλά, καλά. Θα συνεχίσουμε, αλλά θα επιμείνω στα γερμανικά, γιατί και η συνάδελφός μου μίλησε Ιταλικά και Μέχρι τώρα πάντοτε έχει λειτουργήσει το σύστημα, πιστεύω θα λειτουργήσει και σήμερα. 542 στη σελίδα 75 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 545 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και αυτή 548 σε ψηφορία κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα λοιπόν της 548 ψηφίσατε τέλος Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε 549, πρώτο τμήμα πάλι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτό. 546, υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές. Επαλήθευση 546. Ζητώ να αντικατασταθεί ο Ισπανός μεταφραστής. Ισπανός διαρμηνεύσει. Να πει Παρακαλώ να πάρει κάποιος άλλος τη θέση του. δεν είναι δυνατόν. Μέχρι τώρα καλά τα πήγαινε η Ισπανική καμπίνα, κύριε συνάδελφε, και είναι περίεργο ότι από τη στιγμή που ανέλαβα εγώ την διεύθυνση της ε, ψηφοφορία, ξαφνικά κάτι δεν πάει καλά. Ο Πέτερ Λίζε, πρόταση. Βέβαια ο καθένα εδώ μπορεί να μιλεί την γλώσσα του και δεν το αμφισβητώ αυτό. Ο κύριο Ζαλέσκι ωστόσο επεσήμανε κάτι σωστό. Στη γερμανική γλώσσα όταν εκφωνεί κανεί ένα τριψήφιο αριθμό τα δύο τελευταία ψηφία αντιστρέφονται. Θα ήταν πιο εύκολο λοιπόν πράγματι ο πρόεδρος να λέει 5, 4, 8 αντί να λέει 5 και 8 και 4 όπως είναι στα γερμανικά. Καλά λοιπόν, ας προσπαθήσουμε. Νομίζω όμως στην Επιτροπή Περιβάλλοντος έχουμε διεξαγάγει πολλές ψηφοφορίες που πάντοτε πήγανε καλά. Μόνο σήμερα κάτι δεν γίνεται. διακόπτει κάποιος από κάτω. Κύριε συνάδελφε, αν θέλετε αυτοσυγκρατηθείτε λίγο για να προχωρήσουμε. 546, επαλήθευση ηλεκτρονική. Ψηφίσατε. Πέρασε. Απερίφθη. Συνεχίζουμε. 547. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές η ηλεκτρονική επαλήθευση. 5.47. Πέρας. Απερίφθη. Συμβαστική τροπολογία 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται στη σελίδα 78. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Ξαναλέω. 5-5-3. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εκπίπτει το δεύτερο τμήμα. Μήπως μπορείτε να μου το πείτε και με ήπιο τρόπο δεν χρειάζεται να φωνάζετε. Επαληθεύουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα της 553. Ευχαριστώ. Ψηφίσατε. Πέρασε. Απερίφθη. Εκπίπτει το δεύτερο μέρος και συνεχίζουμε με την 562. Υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, δεν ψήφισατε όλοι. Επαλήθευση 562. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. 6 της απασχολήσεως υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 560, 560, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. επαληθευση καλώς, 560 μετά από έτοιμά σας ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. Συνεχίζω. Συμβαστική 38 στην επόμενη σελίδα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πέντε 575 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της ίδιας υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ηλεκτρονική επαλήθευση. Δεύτερο τμήμα της 575. Ψηφίσατε πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 39 και 41 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Συνεχίζω με την σελίδα 84 ή 85, συμβαστική 42, συμβαστική τροπολογία 42, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 601 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 599 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται σύντομη επαλήθευση εδώ μεταξύ μας Πρόεδρος. Τροπολογία 608 ως προσθήκη στην συμβαστική 23. Υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Τέλος. Απερίφθη. 613 ψηφίζουμε τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 614 υπέρ κατά Αποχέσει δεν είναι σαφές η ηλεκτρονική επαλήθευση 614 ψηφίσατε τέλος σαφώς εγκρίνεται 617 και 619 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή εγκρίνονται 616 και 618 είναι ταυτόσιμες και ψηφίζονται μαζί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 620 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 44 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συνεχίζω στη σελίδα 90 στο δικό μου έγγραφο. 637. 637. Σελίδα 90. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Επαλήθευση ωστόσο, 637, η ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει. Ψηφίσατε. Πέρας. Απερίφθη. Συμβαστική 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στη σελίδα 91 τώρα 636 636 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση 636 η ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίσατε πέρας εγκρίνεται λοιπόν 650 εκπίπτει 657 στη σελίδα 92 τη δική μου, συνεχίζω με αυτήν, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Θέλετε επαλήθευση. Καλά λοιπόν, 657 μετά από έτοιμά σας. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. Απερίφθη. 655 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται επαλήθευση 655 αρχίζει ηλεκτρονικά εννοείται ψηφίσατε τέλος απεριφθεί όντως 658 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Η ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 833 είναι η επόμενη. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συνεχίζω σελίδα 94-95 668 668 υπέρ κατά απορρίπτεται 670 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές αυτό απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 51 στη σελίδα 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή συμβαστική τροπολογία μάλλον όχι εμπλόι δηλαδή 15 υπέρ Στη σελίδα 98 για μένα, έμπλου 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε με την συμβαστική 53 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτή. Σελίδα 102 ή 103 Συμβαστική 55 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 576 υπέρ, κατά, τμήμα μόνο των συναδέλφων ψηφίζει διανατάσσεως τη χειρό γι' αυτό ψηφίζουμε ηλεκτρονικά 576. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική τροπολογία 54. Στην επόμενη σελίδα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 736 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 737 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 57 στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Τώρα συνεχίζω στη σελίδα 107 με την 760. 760 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε επαλήθευση. Μάλιστα. Της 760 αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος απερίφθη. 763 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 763 λοιπόν. Ζητείτε επαλήθευση. 763. Οκ. Okay, αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. Απερίφθη. 767 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 768 υπέρ. Ζητείτε επαλήθευση για την 767. Αρχίζει η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 767. Ψηφίσατε. Τέλος. Απερίφθη. 768 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 774 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 779 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 60 υπέρ. Για την 779 θέλετε επαλήθευση. Καλώς. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. Στην σελίδα 110 τώρα, τροπολογία 775. Ψήφι υπέρ, όπως είπα, ψηφίζεται την 775 στη δική μου, στο δικό, μου έγγραφο είναι στη σελίδα 110. Γνωρίζω ότι υπάρχουν και άλλες λίστες ψηφοφορία με διαφορετική αρρύθμιση σελίδων. 775 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα, συνεχίζουμε στη δική μου επόμενη σελίδα με την απασχολήσεως 9, έμπλ 9, δεύτερο τμήμα, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, έμπλ 11, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 784 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συγγνώμη 819 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ηλεκτρονική επαλήθευση 819 λοιπόν τέλος Σαφώς εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 62 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. 434 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ. Καλά λοιπόν. 434 μετά από έτοιμά σας υπέρ. Κατά Μάλλον, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ε, έληξη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Όπως βλέπετε. 435 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 782. Θέλετε παλήθευση για την 435. Ωραία. Αρχίζει. Ηλεκτρονική παλήθευση 435. Ψηφίσατε. Τέλος εγκρίνεται. 782 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση της συμβαστικής 64 αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος εγκρίνεται. Τώρα συμβαστική 64α υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και αυτή. Στη σελίδα 113 τώρα η συμβαστική 63 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα συνεχίζω στην 116 δική μου, σελίδα δηλαδή, με τροπολογία 802 πρώτο τμήμα. Τη βρήκατε, ωραία λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε επαλήθευση. Καλά λοιπόν, 802 πρώτο τμήμα, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. Καλά λοιπόν που κάναμε την επαλήθευση. ...873 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θέλετε τσεκ. 873 λοιπόν επαλήθευση. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται λοιπόν πράγματι. Ακολουθεί 802 τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολία 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση λοιπόν. Συμβαστική 65. Μετά από έτοιμά σας. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται λοιπόν. Και συνεχίζω. Συμβαστική 67 στη σελίδα 118. 67 κατά άποχες εγκρίνεται 807 είναι η επόμενη υπέρ κατά αποχές αυτή απορρίπτεται ακούω έτοιμα; Συγγνώμη, παρακαλώ, να σας διακόψω λίγο. Πρέπει να ψηφίσουμε την συμβαστική τροπολογία 68 ακόμη. Υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Μετά είχατε ζητήσει, μου φάνηκε τσεκ τσεκ τσεκ ότι άκουσα για την 807. Όχι, δεν επιθυμείτε. Καλά λοιπόν, προχωρώ. ...875 στη σελίδα 121. 875. Υπέρ, κατά, αποχές,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 Το δεύτερο τμήμα τώρα της 875 υπέρ, κατά, αποχές δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση 875 δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. 816 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. 832 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 817 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 821 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται λέει ο πρόεδρος, αλλά ακούγονται φωνές για τσεκ. 821 λοιπόν, μετά από έτοιμά σας ηλεκτρονική επαλήθευση 821. Ψηφίσατε. Τέλος. Απορρίπτεται. 844 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική υπαλλήθευση της 844. Ψηφίσατε. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβαστική 69 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 της Επιτροπής Απασχολήσεως υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές. Έμπλ 8 λοιπόν ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. 834 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπολ 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και έμπολ 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή συμβαστική τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και η επόμενη είναι η συμβαστική 72 στη σελίδα 124 ή 25 υπέρ κατά αποχές αυτή απορρίπτεται θέλετε check καλά λοιπόν 72 η ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχισε ψηφίσατε τέλος απορρίπτεται Τότε ακολουθεί 901 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 912 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή. 800 α, θέλετε έλεγχο. Επαλήθευση της 912 μετά από έτοιμά σας. Ψηφίσατε. Πέρας. Απερίφθη. 849 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 849 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται ομοίως. 850 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 798 και 846 είναι ταυτόσιμες και γι' αυτό ψηφίζονται μαζί υπέρ κατά δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ωστόσο οι δύο αυτές 798 και 846 επαληθεύονται ηλεκτρονικά τέλος εγκρίνονται 851 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 852 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ακολουθεί η 859 στην 127 σελίδα 859 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αυτή 862 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 874 η ε, κυρία Χίπνερ ζητεί επαλήθεση της 862 ψηφίσατε όλοι και όλες πέρας απερίφθη κυρία Χίπνερ 874 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Επίσης, συμβαστική τροπολογία 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 864 στη σελίδα 128 ή 29 υπέρ με συγχωρείτε μια στιγμή, μια στιγμή, εδώ υπάρχει μια διαφορά απόψεων. ...876 είναι το σωστό τώρα... ...υπέρ... ...κατά... ...αποχές... ...εγκρίνεται... 879 και 880 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 881 υπέρ. Α. Έτοιμα ηλεκτρονικής επαλήθευσης για τις 79 και 80. Υπέρ. Να μάλλον συγγνώμη. Α, ψηφίσατε όλες και όλοι. Τέλος. Απερίφθη όπως βλέπετε από τα νούμερα. 881 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 882 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 883 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 920 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 884 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία διακόπτει ο πρόεδρος φαίνεται να υπάρχει ένα πρόβλημα με τη γαλλική διερμηνία κύριε Αντελβό συμβαστική τροπολογία 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 890 τώρα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ηλεκτρονική παλιτέψη. 890 πρώτο τμήμα ψηφίσατε πέρας απορρίπτεται και ακολουθεί στην σελίδα 133 στο δικό μου έγγραφο λέει ο πρόεδρος η 896 την βρήκατε ωραία ψηφίπερ κατά αποχές εγκρίνεται 897 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται <coughs> Συμβασική τροπολογία 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μια στιγμή να κάνουμε έναν έλεγχο Wir stimmen DEWE 3. DEWE 3. ΔΕΒΕ 3 ψηφίζεται υπέρ κατά αποχές εδώ θα γίνει επαλήθευση ηλεκτρονική για την ΔΕΒΕ 3 ψηφίσατε τέλος εγκρίνεται 900 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 902 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 903 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 905 905 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα 905 λοιπόν, η ηλεκτρονική επαλήθευση, αρχίζει, ψηφίσατε, τέλος. Εγκρίνεται λοιπόν. Συμβαστική τροπολογία 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση για να είμαστε πιο σίγουροι. Συμβαστική τροπολογία 81 λοιπόν. Ηλεκτρονικά Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε στην σελίδα 134 με ΔΕΒΕ 9 ή 136 του κειμένου του γερμανια DEV DV9 υπέρ, κατά, συγγνώμη, υπέρ ακόμη, κατά, αποχές εγκρίνεται 9-15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9-16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύε 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επαλήθευση μετά από ετοιμά σας. Δεύε 11. Ψηφίσατε. εγκρινεται 9-19. 919. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 914. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 241. Υπέρ. Κατά. Εποχές. απορρίπτεται αυτή. Επαλήθευση του 241 μετά από έτοιμά σας. Ψηφίσατε. Τέλος. Απερίφθη. Η ΤΕΒΕ 12 εκπίπτει και ακολουθεί Τροπολογία 52. Υπέρ. Πρόκειται την αιτιολογική σκέψη α. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τσεκ λοιπόν την 52. Καλά. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. Απερίφθη. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές ασαφές το αποτέλεσμα ηλεκτρονική επαλήθευση 53 Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. 46 έξι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 48 οχτώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική παρήθευση για την 49. Ψηφίσατε. Τέλος. Με μεγάλη πλειοψηφία, μάλιστα, εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Υπέρ λοιπόν. Κατά αποχές εγκρίνεται. 57 δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. 59 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική παρήθευση 59 αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ λοιπόν για την 61 μετά από έτοιμά σας. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται λοιπόν. 56, 60 και 62 όλες μαζί υπέρ κατά αποχές 56, 60 και 62. Στην λίστα μου είναι το λεγόμενο αγγλιστή block vote. Όλες μαζί λοιπόν. Και έτσι θα ψηφιστούν. Η κυρία Ντελβό. Εμείς έχουμε ξεχωριστές εδώ. Φαίνεται πως υπάρχει πρόβλημα που προκύπτει από τις διαφορετικές λίστες ψηφοφοριών των ε, διαφόρων πολιτικών ομάδων. Ωραία. Πολύ καλά λοιπόν. Θα ικανοποιήσουμε το έτοιμά σας ξεχωριστά. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Ε, πλειοψηφία είναι αυτή. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αυτή απερίφθη. Αλλά ας την ελέγξουμε. 62. ηλεκτρονική παλήθευση 62 υπέρ. Συγγνώμη, και ε, ψηφίσατε όλοι, θέλω να πω. Μάλιστα, εγκρίνεται και αυτή λοιπόν. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. αποχέ, εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Α, ε, έτοιμα επαλήθευση της 67. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται λοιπόν. 68 υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές ηλεκτρονική επαλήθευση 68 αρχίζει ψηφίσατε τέλος εγκρίνεται συμβαστική 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές 74 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά 85. Ψηφίσατε. Τέλος. Απερίφθη. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά αποχές αυτή απορρίπτεται τσεκ λοιπόν 89 μετά από έτοιμά σα. ψηφίσατε τέλος απερίφθη 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ τσεκ 86 καλώς λοιπόν αρχίζει η ψηφοφορία ψηφίσατε 86 ηλεκτρονική επαλήθευση τέλος εγκρίνεται λοιπόν 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έτσι είναι ναι επαλήθευση της 92 ψηφίσατε τέλος σαφώς εγκρίνεται Ο 93. 93 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση λοιπόν. Καλά. 93. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται λοιπόν. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ενενήντα πέντε υπέρ κατά απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90, 96 και 97 είναι ταυτόσιμες. Όλες μαζί λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Όμως τις επαληθεύουμε. 90, 96 και 97 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές αυτή εγκρίνεται. Εκατόν εφτά υπέρ. Εμπιστεύομαι τον γραμματέα που μου λέει ότι πρέπει να ψηφιστεί. Στη δική μου λίστα ψηφοφορίας λέει εάν εγκριθεί 100 ή 111 τότε ψηφίζουμε. 107 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 106 εκπίπτει. 101 επίσης. Ψηφίζουμε την 112 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. 112 λοιπόν. Επαλήθευση. Αρχίζει. έληξη τώρα. Εγκρίνεται. Ψηφίζετε την 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. 102 ηλεκτρονική παρήθευση. Ψηφίσατε. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η επόμενη είναι η 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 108 υπέρ εκπίπτει όντως 109 λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 115 υπέρ α ζητείτε επαλήθευση της 114 αρχίζει η ψήφος ψηφίσατε λήξη Με μικρή πλειοψηφία λοιπόν εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πάλι χρειάζεται εδώ ηλεκτρονική επαλήθευση. 115. Ψηφίσατε. Λήξη. Απερίφθη. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ηλεκτρονική επαλήθευση 118 αρχίζει ψηφίσατε λήξη Απερίφθη. Συμβαστική 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ακολουθεί η 129. Στη σελίδα 144. Τη δική μου λέει ο πρόεδρος. 129. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αυτή. 130 υπέρ. Α, θέλετε τσεκ λοιπόν της 129. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Λήξη της ψήφου απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Check this one, λέει η κυρία Τελκαστήγιο. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Λήξεις. Εγκρίνεται. Βλέπετε, λέει η κυρία Τελκαστήγιο. 131. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας γίνει και εδώ η επαλήθευση αρχίζει λήξεις εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα 137 λοιπόν επαλήθευση ψηφίσατε λήξεις απερίφθη 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ζητείτε επαλήθευση αρχίζει ψηφίσατε λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τσεκ καλά λοιπόν 146 μετά από ιδιαίτερο αίτημα ψηφίσατε λήξεις της ψήφου απερίφθη 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 150 υπέρ 150 ηλεκτρονική επαλήθευση. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. 154 λοιπόν ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε. Λήξεις της ψήφου. Απερίφθη. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τσεκ, τσεκ, λέει η κυρία Δελκαστήγιο. 155 μετά από έτοιμά σα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Λήξεις. Απερίφθη. 157 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα 157 ηλεκτρονική υπολήθευση ψηφίσατε λήξη εγκρίνεται 158 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 163 υπέρ κατά εγκρίνεται 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 166 θέλετε επαλήθευση 165 μάλιστα αρχίζει Ψηφίσατε. Λήξεις. Εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 169 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 179 υπέρ κατά αποχές αποτέλεσμα ασαφές Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε. Λήξεις. Εγκρίνεται. 180 υπέρ. Κατά. Πάλι δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. 180 λοιπόν ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Λήξη. Εγκρίνεται. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. 185 λοιπόν ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε. Ξαναλέω, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε. Λήξη. Σαφώς εγκρίνεται. 186 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 189 υπέρ α θέλετε επαλήθευση για την 188 ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίσατε τέλος εγκρίνεται λοιπόν 189 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για, τον κύριο Σεδό ή Αλαμπάρτ, ο οποίος έχει κάτι να ανακοινώσει. Στην τροπολογία υπάρχει ένα σφάλμα, λέει 2013, ενώ το σωστό είναι 2030. Καλώς το ψηφίζουμε τότε το κείμενο με την διόρθωση 2030 και επαναλαμβάνω είναι η τροπολογία 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 191 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές 191 λοιπόν ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίσατε λήξη σαφής έγκριση. 193 λοιπόν υπέρ κατά αποχές δεν είναι καθόλου σαφές το αποτέλεσμα 193 ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίσατε τέλος εγκρίνεται 194 υπέρ κατά αποχές αυτή απορρίπτεται. Επαλήθευση λοιπόν, καλά, 194 μετά από έτοιμά σα ψηφίσατε, λήξη, απερίφθη. 195 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 196 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 197 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 199 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 204 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 208 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. υπαριθμών 1 αλλά και μέχρι 4 όλες μαζί. 1, 2, 3, 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση. Καλά. Τροπολογία 5. Ψηφίσατε. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται πράγματι. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Υπαριθμών 7, 9, 11 και 10 όλες μαζί. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Προπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 και 15 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 16, 17, 18 πάλι όλες μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Αν θέλετε τσεκ, πριν από το τσοκ, 16, 17, 18 όλες μαζί. Ψηφίσατε. Λήξη. Εγκρίνονται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 και 21 μαζί. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 23, 24, 25 και 26 πάλι αυτές όλες μαζί, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Ακολουθούν 28 και 30 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. πάλι όλες μαζί. 32, 35, 36, μέχρι 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τώρα 33. 33. που είναι στην σελίδα 153. 33 ξαναλέω, υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι το αποτέλεσμα, ηλεκτρονική παρήθευση 33. Ψηφίσατε. Λήξη. Εγκρίνεται λοιπόν. 34 υπέρ κατά αποχές οι σοσιαλιστές δεν σηκώνουν πια τα χέρια οι 34 ψηφίστε ξεχωριστά λέει ο πρόεδρος υπέρ λοιπόν κατά αποχές απορρίπτεται λοιπόν αυτή 38. Α, ζητείτε τώρα τσεκ του 34. Καλά λοιπόν, αρχίζουμε. Ψηφίσατε. Λήξεις. Απερίφθη. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ομοίως. μια στιγμή να βεβαιωθούμε ότι δεν έχουμε κάνει κανένα λάθος. Από την ε, ομάδα των φιλελευθέρων έχει ζητηθεί διακοπή για λίγα λεπτά. Αρχικά έτσι είχατε πει. Ο κ. Ντέιβις. Πράγματι είχα ζητήσει να υπάρξει ένα διάλειμμα πέντε λεπτών η αίσθησή μου είναι ότι τώρα διαμορφώθηκαν τα πράγματα και οι αντιλήψεις για το πώς θα ψηφίσουν δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει τέτοια διακοπή. Σαν συνεισηγητής για τη συγκεκριμένη έκθεση θα ήθελα να ενθαρρύνω όλα τα μέλη ...τη ΣΥΤΡΕ και της Επιτροπής Επισπεριβάλλοντος να καταψηφίσουν. Για ένα απλό λόγο. Εκτιμώ βέβαια ότι εμείς θα μπορούσαμε να δεχθούμε τις πιο ριζοσπαστικές προτάσεις για μειώσεις των εκπομπών. Αλλά ο τριπλασιασμός των στόχων δείχνει ότι δεν καταλάβαμε τα μαθήματα του παρελθόντος και δεν δίδουμε τις σωστές απαντήσεις για τις οικονομικές ευρωπαϊκές προκλήσεις. Υπήρξατε σαφής, λέει ο Πρόεδρος. Θα ψηφίσουμε. Δεν υπάρχουν προσωπικές τοποθετήσεις. Έχετε να πει κάτι επί της διαδικασίας. Ε, κύριε Τερκαστήγιο. Κοιτάξτε, είχαν ε, ζητηθεί κάποια λεπτά και εγώ είχα ζητήσει δύο-τρία λεπτά γιατί χρειάζεται να μιλήσω με τα μέλη της πολιτικής μου ομάδας. Είναι χρήσιμο να γίνει κάτι τέτοιο, ήταν πολύ περίπλοκη η ψηφοφορία και απαιτείται να έχουμε δύο-τρία λεπτά στη διάθεσή μας. Ο συνάδελφος Κριστέιβης απέσυρε το αίτημά του και από ό,τι βλέπω η κυρία Καστίγιο θέτει τώρα αίτημα διακοπής λίγο, λίγων λεπτών. Στις 11 και 40. Στις 11 και 40 λοιπόν ψηφίζουμε, ε, κάνουμε την τελική ψηφοφορία.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 Παρακαλώ όλες και όλους τους συναδέλφους καθώς και τους διαφόρους επισκέπτας. Ησυχία παρακαλώ για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ευθύς αμέσως με την πρέπουσα τάξη στην τελική ψηφοφορία. Όλα τα μέλη είναι πάλι εδώ και ψηφίζουμε τώρα σε τελική ψηφοφορία, βεβαίως ηλεκτρονικά αρχίζει η τελική ψηφοφορία της εκθέσεως. Ψηφίσατε, όλες και όλοι ψηφίσατε. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε η έκθεση με 66 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 3 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια και στον εισηγητή και ευχαριστώ και την συνάδελφό μου κυρία Σαρτόρη καθώς και τις δύο γραμματείες των Επιτροπών για αυτό το γιγάντιο έργο Λίγη η συνεδρίαση. Παραλίγο να αρχίσω να συνηθίζω αυτή τη συνεργασία μαζί σας κύριε Σαρτόρη.